Επίτροπο Όρμπαν. Τέλος της συζήτησης και θα ψηφίσουμε αμέσως. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στις επεξηγήσεις ψήφου και κατά την διαδικασία Catch the Eye εξαντλήσαμε την διαδικασία αυτή. Πλέον δεν μπορώ να δεχτώ άλλες αιτήσει. από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθείτε. Σύμφωνα με το επόμενο σημείο της μερικής διάταξης έχουμε την ψηφοφορία των έξι ψηφισμάτων, σχεδίων ψηφισμάτων για την Γουινέα. Θα ξεκινήσουμε με την κοινή ψηφοφορία των έξι ομάδων, σημείο 10, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. 73 ψήφισαν, 33 υπέρ, 34 κατά, 6 αποχές απορρίπτεται. Ναι, κύριε Χίγγιν, ζητάτε το λόγο. Πρόεδρε, δεν έχω την κάρτα μου, αλλά θα ήθελα να ψηφίσω υπέρ. Το σημειώνουμε. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα στο αποτέλεσμα. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο? Διαδικαστικό. Και εγώ δεν έχω την κάρτα μου. Και εγώ θέλω να ψηφίσω κατά, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, τα σημειώνουμε όλα αυτά και αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες ε, περιπτώσεις θα πρέπει να τις ανακοινώσετε. Και τώρα ψηφίζουν το, την τροπολογία 1 αναθεωρημένη της ομάδας Άλντε και Πρασίνων. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 74 ψήφισαν, 32 υπέρ, 37 κατά και 5 αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 74 ψήφισαν. Κανείς δεν απέχει, κανείς δεν ψηφίζει κατά. Ομόφωνα εγκρίνεται το ψήφισμα. Αντικαθιστά λοιπόν το παλιό κείμενο. Και τώρα Περνάμε στο κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων για το Ιράν. Ψηφίζουμε το 8 με ξεχωριστή ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και όλα τα υπόλοιπα ψηφίσματα καταπίπτουν και αντικαθιστώνται από αυτό και τώρα περνάμε στην Στριλάνκα. Έξι σχέδια ψηφίσματος, ψηφίζουμε για το κοινό ψήφισμα το οποίο θα αντικαταστήσει τα προηγούμενα. Ψηφίζουμε λοιπόν το σημείο 1, τροπολογία 1 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 2 για το 8 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία και ψηφίζουμε στο 11 την τροπολογία 3 των πρασίνων Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία. Στην τρίτη αιτιολογική σκέψη θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάν που θέλει να κάνει μια προφορική τροπολογία. Προτείνω στο σημείο 3 εδώ να το βγάλουμε τελείως από το κείμενο γιατί όπως ξέρετε ο δημοσιογράφος αυτός δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η ε, κατάστασή του. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, στην τρίτη ε, αιτιολογική σκέψη ζητάτε να μην υπάρξει αυτή η τροπολογία, να το σβήσουμε δηλαδή τελείως το κείμενο αυτό. Εσείς, όχι τότε ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή. Να σβηστεί τελείως η τρίτη ιδεολογική σκέψη. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία του κυρίου Μάν. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 63, 60 υπέρ, 3 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το ψήφισμα. Φτάσαμε και στο τέλος των ψηφοφοριών. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι το ΕΛΚ ζήτησε ο κύριος Γκέρι να γίνει μέλος της ειδική Επιτροπής για την Οικονομική Κρίση. Νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε αυτόν τον διορισμό. Ο κύριος Πόσελ ζητάει το λόγο.